Αγαπητέ Αντιπρόεδρε, εξοχότατη, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι. Είναι μέγα προνόμιο για μένα η ευκαιρία που έχω να καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον κύριο Τζόζεφ Μπάιντεν, 47ο Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο αντιπρόεδρος Biden διαδραμάτισε ε, ρόλο κλειδί στην αμερικανική πολιτική και είναι φίλος ε, συναδέλφων και του Κοινοβουλίου εδώ και χρόνια. Το 1972 εξελέγει για πρώτη φορά γερουσιαστής. Ε, ήταν ένας από τους νεοτέρους τότε γερουσιαστές στην ιστορία της χώρας. Επανεξελέγει έξι φορές πριν ε, ε, γίνει αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να κλεγεί το Νοέμβριο του 2008. Πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Γερουσίας και της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Είναι γνωστός για τον ευθύ του λόγο, την ειλικρίνειά του και πολλές φορές για θέματα που δεν είναι δημοφιλή. Καθοδηγεί την κοινή γνώμη, δεν την ακολουθεί. Γι' αυτό και σήμερα η μιλία σα, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τόσο σημαντική, τόσο κρίσιμη για όλους μας. Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω και πάλι για την θερμότατη σας πρόσκληση και την τόσο επικοδομητική και καρποφόρα συζήτηση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον. Αγαπητοί συνάδελφοι, στο σημερινό κόσμο που είναι πολυμερής και πολυπολικός, η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να συνεργάζονται σε εταιρική σχέση για την παγκόσμια σταθερότητα και για τις πεφωτισμένες αξίες τις οποίες πιστεύουμε. Η επίσκεψη του Προέδρου Biden σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδεικνύει ακριβώς αυτή τη δέσμευσή μας. Χρειάζεται ισχυρή και αποτελεσματική ε, διατλαντική εταιρική σχέση, επίσης όρη. Άλλω, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρώπη δεν μπορούμε να βρούμε βιώσιμε λύσει σε πολλέ προκλήσει που αντιμετωπίζουμε. Ενεργειακή ασφάλεια, οικονομική κρίση, κλιματική αλλαγή. Είναι ε, θέματα που μα πλήττουν ακόμα όλου ακόμα η καταπολέμηση τρομοκρατίας, η προώθηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων, η περάσπιση του ελευθερού εμπορίου και η παγκόσμια διακυβέρνηση. Πριν από 25 χρόνια, αγαπητοί συνάδελφοι, περίπου μέρα, την ίδια μέρα, ο πρόεδρος Ρέγκαν στις 8 Μαΐου ε, το 1985 μίλησε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν η τελευταία ε, φορά που ένας Αμερικανός πρόεδρος και μοναδική μίλησε ενώπιον ε, κλεγμένων προσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η παρουσία σας σήμερα εδώ κύριε Αντιπρόεδρε ε, σηματοδοτεί την επανάληψη αυτού του διαλόγου σε ε, υψηλότερο επίπεδο μεταξύ των δύο πύρων. Στην Ευρώπη σήμερα έχουμε μια νέα συνθήκη, είναι και πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εμά νέα ισχύ, ε, νέα δυνατότητα δράση. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι ΔΕ Ηνωμένε μετά από ένα χρόνο ε, ηγεσία του Προέδρου Ομπάμα, διαγράφεται μια νέα ελπίδα για τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη η επίσκεψή σας κύριε ε, Αντιπρόεδρε. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Κοινοβούλιο της Ευρώπης και έχετε το λόγο. Mr. President, thank you for that welcome. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για αυτή την, το, αυτό το καλωσόρισμα. Ήταν μεγάλη χαρά να σας έχουμε στη Washington στο Λευκό Οίκο και είναι μεγάλη τιμή. Μπορώ να πω και προνόμιο το να βρίσκομαι ενώπιον αυτού του διακεκριμένου σώματος. Εγώ υπηρέτησα σε ένα κοινοβούλιο που είχε μόνο 435 μέλη. Εδώ είναι ακόμα μεγαλύτερη η τιμή που νιώθω. Θυμάμαι τον λόγο του Προέδρου Ρέγκαν εδώ το 1985 και για να παραθέσω τον ε, William Butler Yeats, που, τον Ιρλανδό ποιητή, που σε ένα ποίημα που λεγόταν ε, Πάσχα του 1969, οι στίχοι του έλεγαν «Όλα έχουν αλλάξει, Μία τρομερή ομορφιά έχει δημιουργηθεί. Πολλά έχουν ε, αλλάξει από το 1985 και μια τρομερή ομορφιά έχει όντως γεννηθεί. Και όπως ήδη γνωρίζετε κυρίες και κύριοι, είμαι Ευτυχή που βρίσκομαι στι Βρυξέλλε για δεύτερη φορά ω αντιπρόεδρος και όπως πιθανότατα θα γνωρίζετε ορισμένοι πολιτικοί και αμερικανοί δημοσιογράφοι αναφέροντας την Washington DC ως ε, την πρωτεύουσα του ελεύθερου κόσμου. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτήν εδώ την ε, σπουδαία πόλη που έχει χίλια χρόνια ιστορία και που είναι πρωτεύουσα του Βελγίου αλλά και πρωτεύουσα ολόκληρης Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στρατηγείο του ΝΑΤΟ έχει τη δική τη ξεχωριστή αξία ε, Έχω υπηρετήσει για πάνω από 36 χρόνια στο δικό μας ε, κοινοβούλιο και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που μπορώ σήμερα να απευθυνθώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος ε, Ομπάμα ο πρώτος έγχρωμος πρόεδρος που ανέλαβε τα καθήκοντα πρόεδρου στην Αμερική Πραγματικά ε, έχει σημάνει διαφορά και, και ο ίδιος εκφράσει τη μεγάλη του εκτίμηση για τη δουλειά που κάνετε εσείς εδώ στο... στο προπύργιο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Εσείς αντιπροσωπεύετε 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Σκεφτείτε δύο εκλεγμένα σώματα που νομοθετούν για το ένα οδό του πληθυσμού ολόκληρου του πλανήτη. Αυτό είναι πολύ εξωσημείωτο και τώρα με την συνθήκη της Λισαβόνας έχετε αναλάβει περισσότερες εξουσίες και μεγαλύτερες ευθύνες που συνοδεύουν αυτή την αυξημένη επιρροή. Και αυτό το καλωσορίζουμε. Το καλωσορίζουμε γιατί εμείς οι ΙΠΑ χρειαζόμαστε ισχυρούς συμμάχους και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του 21ου αιώνα. Πολύ... Πολλά είναι ταυτόσημα, αλλά όχι διαφορετικά από τον προηγούμενο αιώνα. Για να τα αναφέρω. Η κυβερνηση ομπαμα Ομπάμα-Μπάιντεν δεν έχει καμία αμφιβολία όσον αφορά την ανάγκη για ισχυρή στήριξη μιας ζωντανής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύουμε πως είναι απολύτως απαραίτητο για την Αμερικανική ευημερία και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Να μην έχετε καμία αμφιβολία περί αυτού. Όταν ε, προείδρευσα τις ε, Επιτροπή τη Γερουσία για τις Εξωτερικές Επιθέσεις για πολλά χρόνια είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με πολλούς ε, από εσά που είστε εδώ μέσω των Εθνικών Κοινοβουλίων και των ε, Εθνικών Επιτροπών ε, εξωτερικών υποθέσεων. Εκτιμώ πόσο δύσκολο ήταν να οικοδομηθεί το μόνο πολυεθνικό κοινοβούλιο του κόσμου που εκλέγεται με καθολική ψηφοφορία. Τόσα πολλά έχουν αλλάξει και είμαι πολύ ευχαριστημένος που μέσω της, ε, του διαλόγου του διατλαντικού μεταξύ των νομοθετών δημιουργείται μια στενή σχέση ανάμεσα σε εσά και το Κογκρέσο και ελπίζω πως η επαφή ε, της του περασμένου μήνα στη Washington θα βελτιώσει ακόμη περισσότερο αυτούς τους δεσμούς. 65 χρόνια... 65 ε, χρόνια πριν οι ηγέτες των Ναζί ε, λίγο νοτιότερα από εδώ υπέγραψαν ε, την, ε, την, την παράδοσή τους ανεφόρων. Κόσμος επεφημούσε σε ολόκληρη τη Σαν Ζελιζέ και σε ολόκληρο τον κόσμο και εδώ στις Βρυξέλλες έγινε μια λειτουργία ευχαριστειών ακούστηκαν οι εθνικοί ύμνοι του Βελγίου, της Βρετανίας, των Ηνωμένων Πολιτειών σε εκείνη την ωραία μέρα, 8 Μαΐου 1945, αυτή η Ήπειρος ε, ήταν ε, ρήπια. Είχε ε, καταρακωθεί από δύο παγκοσμίους πολέμους σε λιγότερο από 30 χρόνια. Και εκείνη τη στιγμή μια Ευρώπη ειρηνική, ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα φαινόταν σαν όνειρο για οποιονδήποτε. Κι όμως, μέσω της βούλησης των συμπολιτών σας και πολιτικών ανδρών όπως ο Πόλαν Ρισπάκ, ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Ζαμόνε, οραματιστές που έδωσαν ζωή σε ένα κοινοβούλιο και ε, ε, προχώρησαν με βάση το προεδρικό μοντέλο του Λίντον Τζόνσον να είμαστε εδώ, να είστε εσείς εδώ. Αυτό που ξεκίνησε με 5-6 κράτη, με την ΕΚΑΧ, μόνο με την κοινή αγορά άνθρακα και χάλιβα, σε, οδηγήθηκε σε μια κοινότητα που είναι αφοσιωμένη στην ελεύθερη σκέψη, την ελεύθερη κίνηση και, την και το ελεύθερο εμπόριο. Την ελεύθερη Ευρώπη, που δεν είναι μόνο ένας χώρος, αλλά είναι μια ιδέα, ένα ιδανικό. Και εγώ εδώ αντιπροσωπεύω τον πρόεδρο Ομπάμα και πιστεύω σε αυτή την ιδέα και σε ένα καλύτερο κόσμο, μια καλύτερη Ευρώπη, που ήδη, έχουν βοηθεί, που, που ήδη έχει δημιουργηθεί. Μια Ευρώπη όπου όλα τα κράτη-μέλη θα χαίρουν μέσω της διαπραγμάτευσης εμπορικών συμφωνιών και μέσω της αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών με μια ενωμένη φωνή. Μια Ευρώπη που υποστηρίζει τις ε, πολιτικές και πολιτιστικές αξίες τις οποίες συμμερίζεται η χώρα μου ε, μαζί σας. Μια Ευρώπη ολόκληρη, ελεύθερη και ειρηνική. Όπως είπε ο πρόεδρος Ομπάμα στην Πράγα πριν από ένα χρόνο μόλις, σε μια, ενισχυ... μια ισχυρότερη Ευρώπη σημαίνει ισχυρότερο εταίρο για τις ε, ΗΠΑ και χρειαζόμαστε ισχυρότερους εταίρους και γι' αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε αυτή την τεράστια προσπάθειά σας. Για τα περασμένα 65 χρόνια μας έδειξαν ότι όταν οι Αμερικανοί και η Ευρώπη αφιερώνουν την ενέργειά τους σε κοινού στόχους, δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να μην μπορούν να καταφέρουν. Μαζί με το σχέδιο Μάρσαλ αν, ε, ολόκληρη την Ευρώπη. Μαζί φτιάξαμε την πιο μόνιμη συμμαχία ασφάλειας στο ΝΑΤΟ και την μόνη πολιτική μια δύναμη που μας φέρνει κοντά Αμερικανούς και Ευρωπαίους τα τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε φτιάξει, έχουμε θεσπίσει τις πιο αρμονικές εμπορικές σχέσεις στην ιστορία του κόσμου. 40% των συναλλαγών έχουν επιφέρει άνευ προηγουμένου ευημερία και τεχνολογική πρόοδο. Μαζί παρέχουμε ανακούφιση και ελπίδα για όλο τον κόσμο που υποφέρει από τα Δυτικά Βαλκάνια μέχρι το Κονγκό, μέχρι τη λεγόμενη δουλειά μας στην IT σήμερα. Σε όσους σκεπτικιστές που παρά όλα αυτά τα επιτεύγματα εξακολουθούν να πιστεύουν και να αμφισβητούν την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων και, τις, ε, και έχουν αμφιβολίες για τις σχέσεις μεταξύ ΙΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σας πω το εξή. Ακόμα και αν η ΙΠΑ και τα κράτη τα οποία εσείς αντιπροσωπεύετε δεν ενώνονταν από κοινό πολιτισμό και κοινέ αξίες πολλών εκατομμυρίων πολιτών μας και μόνο και μόνο τα παγκόσμια μας συμφέροντα θα μας έδαιναν μεταξύ μας. Οι σχέσεις μεταξύ της χώρας μου και της Ευρώπης είναι σήμερα τόσο δυνατή και τόσο σημαντική όσο ήταν ποτέ. Αυτό ο αιώνας έχει ε, απελευθερώσει, έχει μάλλον οδηγήσει σε νέες προκλήσεις και μαζί τις αντιμετωπίζουμε μία προς μία. Είναι δύσκολες, θα υπάρξουν διαφωνίες, αλλά τις αντιμετωπίζουμε κοινά. Κλιματικές αλλαγές, μια από τις μεγαλύτερες απειλές που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας. Η και η Ευρώπη συνεργάζονται ώστε να εξασφαλίσουν ότι όλες οι χώρες και κυρίως οι μεγάλες οικονομίες θα συμβάλλουν για μια παγκόσμια λύση. Όλοι προσβλέπουμε και κάναμε σημαντικά βήματα μπροστά στην Κοπενχάγη. Τώρα θα πρέπει όλες αυτές τις περικοπές στις εκπομπές να τις υλοποιήσουμε και να χρηματοδοτήσουμε τη διαφάνεια την οποία ζητάμε σε αυτή τη συμφωνία. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε τις πιο ευάλωτες χώρες από τον Αρκτικό Βορρά μέχρι τα νησιά του Ειρηνικού πέρα από το τοπίο του Αφγανιστάν και του Πακιστάν συνεργαζόμαστε για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο από τους Ταλιμπάν αλλά και να εκπαιδεύσουμε μια στρατιωτική και αστυνομική δύναμη στο Αφγανιστάν ώστε να μπορεί να προστατεύσει τον ίδιο το λαό να μπορέσουμε να φτιάξουμε κυβερνητικές δυνατότητες εκεί στο Αφγανιστάν. Η Αμερική και η Ένωση αφιερώνουν σημαντικούς στρατιωτικούς και πολιτικούς πόρους για να συντηρήσουν αυτές τις σημαντικές ε, αποστολές. Πράγμα που δεν είναι πάντα πολύ δημοφιλέ, αλλά γνωρίζετε όλοι πω χρειάζεται. Και ω ηγέτε είμαστε υποχρεωμένοι να αποδείξουμε στου πληθυσμού μα ότι αυτό είναι απαραίτητο για τη συλλογική μα ασφάλεια. Αν και πιστέψτε μου ε, ότι ω πολιτικό που υπηρετεί εδώ και 30 χρόνια δεν, καταλαβαίνω πως δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν είναι καθόλου δημοφιλές ούτε και στη δική μου χώρα όπως δεν είναι και εδώ. Επίσης, γι' αυτό το λόγο, είναι άλλος ένας λόγος που η Αμερική και η Ευρώπη στέκονται ε, χέρι με χέρι για να εμποδίσουν την εξάπλωση των πυρηνικών όπλων ε, σε χώρες ε, που είναι στενή μα σύμμαχοι. Μαζί ξεκινήσαμε ένα άνευ προηγουμένου δρόμο για αντιμετώπιση ειρηνική των Ιρανών ηγετών. Παρά αυτά που σκέφτονταν ορισμένοι σκεπτικιστές, ο πρόεδρος είπε ότι θα απλώσουμε το χέρι μα σε οποιοδήποτε ε, εταίρο που άνοιγε το χέρι του, που χαλάρωνε τη γροθιά του. Η, η αμερικανική κυβέρνηση Ομπάμα ξεκίνησε με αυτό το πνεύμα, να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη στη διεθνή κοινότητα συμπεριλαμβάνουν χορηγώντας πρόσβαση στους, στις πρώην ε, αδήλωτες εγκαταστάσεις αλλά και επιτρέποντας τη χρήση ενός αντιδραστήρα για την παραγωγή καυσίμου. Ολόκληρος ο κόσμος είδε πως οι Ιρανοί ηγέτες αγνοούν την καλή μας βούληση και συνεχίζουν να προβαίνουν σε ενέργειες που απειλούν τη συλλογική μας σταθερότητα. Όταν μια χώρα παραβιάζει τις υποχρεώσεις της ενάντια στην ε, Διεθνή Συνθήκη για τη Μη Εξάπλωση των Πυρηνικών Όπλων και θέτει σε κίνδυνο μια τεράστια έκρηξη στην ε, Μέση Ανατολή δεν θα ήταν πραγματικά ηρωνικό αφού κατέπεσε το σιδηρούν παραπέτασμα και έχει μειωθεί η απειλή για αμοιβαία καταστροφή ανάμεσα στις υπερδυνάμεις να έρθει και να ξεκινήσει μια νέα, ένας νέας αγώνας εξοπλισμών σε ένα από το πιο ασταθή μέρη του κόσμου. Δεν θα ήταν ηρωνικό πραγματικά τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και τα δυσέγγονά μας ε, να μην μας συγχωρήσουν ποτέ για το τι κάναμε εμείς στο παρελθόν. Επιπλέον, οι Ιρανοί ηγέτες υποστηρίζουν τρομοκρατικές ε, οργανώσεις και χωρίς καθόλου να ντρέπονται διώκουν τους ίδιους τους πολίτες οι οποίοι υποστηρίζουν τη δικαιοσύνη και σύμφωνα με το απιστεύω των δικών μας κυβερνήσεων. Το Ιράν αντιμετωπίζει μια επιλογή. Είτε να έρθει στην κοινότητα των υπευθύνων κρατών, πράγμα που το ελπίζουμε, είτε να αντιμετωπίσει περαιτέρω συνέπειες και αυξανόμενη απομόνωση υπό το φως ε, της απειλής που κρέμεται πάνω από το Ιράν Όλοι φοβόμαστε για την ασφάλεια των ε, συμμάχων μας. Γι' αυτό και αναπτύξαμε το πρόγραμμα πυραυλικής άμυνας σε αυτήν εδώ την Ήπειρο. We're also working together inside NATO. Γι' αυτό και δουλεύουμε μέσα στο ΝΑΤΟ για να καλύψουμε τις μελλοντικές απειλές όπως οι κυβερνοαπειλές, η κυβερνοασφάλεια. Προσπαθούμε να προωθήσουμε διαρκώς όλο και περισσότερο τη στενή συνεργασία μεταξύ ΝΑΤΟ και Ένωσης. Γρήγορα και αποφασιστικά ε, ε, ενεργήσαμε τη στιγμή που απειληθήκαμε από μια οικονομική κρίση πολύ μεγαλύτερη από αυτή της ε, του, κράχ. Παρακολουθούμε πολύ στενά όλη την διάρκεια της κρίσης, τις οικονομικές προσπάθειες, τις προσπάθειες της Ελλάδας και υποστηρίζουμε, καλωσορίζουμε το πακέτο στήριξης που εξετάζει η Ευρώπη στη συνεργασία με το ΔΝΤ και θα το υποστηρίξουμε και θα παρακολουθούμε τις προσπάθειες διάσωσης της Ελλάδας. Αυτά τα παραδείγματα και πολλά άλλα που μπορώ να αναφέρω δείχνουν γιατί η Ευρώπη εξακολουθεί όχι μόνο να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ένωσης αλλά και ο μεγαλύτερος της σύμμαχος. Κυρίες και κύριοι, οι προκάτοχοί μας συγκεντρώθηκαν πριν από 60 χρόνια για να εξασφαλίσουν ότι τα σκοτεινότερα κεφάλαια του 20ου αιώνα δεν θα συνεχίζονταν και στον 21ο. Αυτά τα θεσμικά όργανα ε, ε, αποτέλεσαν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά τώρα θα πρέπει να στραφούμε στις προκλήσεις αυτού του νέου αιώνα που ανέφερα και, στο, και στην αρχή. Ο κόσμος έχει αλλάξει, έχει αλλάξει ρηξικέλευθα μια τρομερή ομορφιά έχει γεννηθεί και ίσως η πιο περίπλοκη ε, πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτή που αντιμετωπίζουμε από τους ίδιους μας τους πολίτες. Δηλαδή όχι από κρατικούς φορείς, ας πούμε αυτούς τους εξτρεμιστές που θέλουν να απλώσουν το χέρι σε οποιοδήποτε όπλο μαζικής καταστροφής. Και ο φόβος, η απειλή δεν έχει σύνορα. Κανένα σύνορο, κανένα κράτος μόνος του, όσο δυνατό και όσο οργανωμένο να είναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους απειλές. Μπορεί να επιτύχει μόνο στο να το περιορίσει αν ε, ε, ε, συνεργαστεί και ακριβώς αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και η συνθήκη της Λισαβόνα σας δίνει μεγαλύτερο ρόλο, μεγαλύτερο ρόλο και πιο υπεύθυνη διακυβέρνηση το Κογκρέσο και το Κοινοβούλιο διαρκώς προσπαθούν να δουν πώς θα προστατέψουν καλύτερα τους λαούς αυτούς όλους. Και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι οφείλουμε και μπορούμε να προστατέψουμε τους πολίτες μας και να διατηρήσουμε τις ελευθερίες μας. Από πέρσι που ανέλαβε, που ανέλαβαμε την εξουσία ο πρόεδρος Ομπάμα και εγώ, έχουμε υπακούσει στην συνταγματική μας επιταγή να επιζητήσουμε μια τελειότερη ένωση. Ε, μια από τις πρώτες επίσημες δράσεις μας ήταν να σταματήσουμε, να απαγορεύσουμε ανακριτικές πρακτικές οι οποίες απέδιδαν λίγα και που δεν μπορούσαμε να τις συνεχίσουμε με ήσυχη συνείδηση. Διατάξαμε το κλείσιμο του κρατητήριου του Γκαντάναμο Μπέι που είχε γίνει σύμβολο αδικίας και σύνθημα των τρομοκρατών. Εκτιμούμε δε ιδιαίτερα την υποστήριξη δύσκολη απόφαση για σας, αλλά τόσο πολύ μας υποστηρίξατε στην προσπάθεια αυτή. Τα κάναμε τα πράγματα αυτά διότι όπως και εσείς, ο πρόεδρος Ομπάμα και εγώ απορρίπτουμε το ψευδοδήλημα ανάμεσα στην ασφάλειά μας και στα ιδεώδη μας θεωρούμε ότι η διατήρηση των ιδεωδών μας μας κάνει πιο ισχυρούς και ότι οποιαδήποτε υπονόμευσή τους υπονομεύει στην πραγματικότητα τις προσπάθειές μας στον ευρύτερο αγώνα κατά της βίας τρομοκρατίας. Ποιος είναι ο στόχος? Ο στόχος είναι να αλλάξουν, αυτό ο στόχος τους, να αλλάξουν αυτά που θεωρούμε εμείς αξίες, να αλλάξουν τους τρόπους συμπεριφοράς μας. Οχτώ μόλις ημέρες μετά από την 11η Σεπτεμβρίου είπα σε χιλιάδες ε, σε μια ομάδα χιλιάδων φοιτητών στην χώρα μου ότι δεν επιτρέπεται να αφήσουμε την τραγωδία της 11 η Σεπτεμβρίου να αλλάξει τον τρόπο ζωής μας, διότι αυτό επιδιώκουν οι τρομοκράτες. Τους είπα ακόμη ότι η Αμερική δεν θα μπορέσει να κατησχίσει στον αγώνα αυτό δρώντας μόνη της. Αυτά τα λόγια μου δεν ανταποκρίνονταν μόνο στο πνεύμα εκείνης της εποχής, αποδείχθηκαν εν τέλει να είναι αλήθεια και είναι ασφαλώς αλήθεια και σήμερα. Δεν χρειάζεται να σας πω σε εσά σχετικά με την ε, υπερήφανη ε, παράδοση που έχετε εδώ προστασίας των πολιτών σας απέναντι σε κυβερνητικές διεισδύσεις στην ιδιωτική τους σφαίρα. Αυτά τα πράγματα είναι αναπαλωτρίωτα δικαιώματα. Το ίδιο βαθιά είναι η δέσμευση της Αμερικής για την προστασία της ιδιωτικής σφαίρας. Το ίδιο βαθιά όπως και εσείς. Η τέταρτη τροπολογία του συντάγματό μα προστατεύει τα άτομα απέναντι σε οποιασδήποτε αδικαιολόγητε έρευνε ή ε, κατασχέσει από το κράτο, κάτι που ορισμένοι από του πιο διάσημους νομικού μα ονόμασαν το δικαίωμα να σε αφήνουν ήσυχο. Το ανώτατο Αμερικανικό Δικαστήριο είπε ότι η ιδιωτική σφαίρα προστατεύεται συνταγματικά και είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Και όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι το ανώτατο συνταγματικό μας δικαστήριο χαρακτήρισε το δικαίωμα αυτό ως θέμα προσωπικής ατομικής αξιοπρέπειας. Τώρα, ε, προσωπικά εγώ για 36 χρόνια στη σταδιοδρομία μου υποστήριξα τα δικαιώματα στην ιδιωτική σφαίρα. Στην Αμερικανική Γερουσία κάθε χρόνο οργανώσεις οι οποίες προστατεύουν την ε, προσωπική σφαίρα και κάθε χρόνο και εγώ και ο πρόεδρος Ομπάμα χαρακτηριστήκαμε σαν από τα πιο σημαντικά πρόσωπα που ε, φροντίζουμε για την προστασία αυτή. Να αλλάξουμε τώρα θα σήμαινε ότι διαψεύδω οτιδήποτε υποστήριξα μέχρι τώρα στην χώρα μου για τα τελευταία 37 χρόνια. Όταν ε, ήμουν πρόεδρος της ε, Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της Γερουσίας που προτείνει και τους υποψηφίους για τις θέσεις δικαστών. Εγώ τους άκουγα πριν να ε, αποφασίσουμε αν θα μπορέσουν να προχωρήσουν για να εκλεγούν στα ε, αξιώματα αυτά. Θεωρεί και ο ίδιος ο πρόεδρος Ομπάμα ως πρώτη στο καθήκον του την προστασία της προσωπικής σφαίρας των πολιτών που εκπροσωπεί. Ο πρόεδρος Ομπάμα είπε ωστόσο ότι η ασφάλεια της πατρίδας είναι το πρώτο πράγμα που τον απασχολεί μόλις ξυπνήσει το πρωί και το τελευταίο πράγμα πριν να ε, ξαπλώσει την κλίνη το βράδυ. Και νομίζω ότι όλοι οι ηγέτες το ίδιο θα πούν. Πράγματι, η προσωπική ασφάλεια του καθενός είναι επίσης αναπαλωτρίο το δικαίωμα όπως και η προσωπική σφαίρα. Η σωματική ακαιρότητα και ασφάλεια είναι επίσης λοιπόν το δικαίωμα. Οποιαδήποτε κυβέρνηση παρετείται από το δικαίωμα να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών της παραβιάζει τα δικαιώματά του. Το ίδιο όπως μια κυβέρνηση η οποία επιβάλλει τη σιγή στους αντιφρονούντες. Και όπως είμαστε εδώ σήμερα και μιλούμε, οι εχθροί μας κάνουν κάθε τι που μπορούν για να ε, προχωρήσουν σε δολοφονικέ απόπειρε όπως αυτές που έπληξαν τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και τη Μαδρίτη. Για να το σταματήσουμε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε προστάσιο διαθέτουμε. Την επιβολή της τάξεω, τη στρατιωτική επιλογή, την συλλογή προφοριών, την τεχνολογία. Αγωνιζόμαστε σε πολλά μέτωπα από του ε, ανδρείους στρατιώτες μας, αμφωτέρων των φίλων βεβαίω που αγωνίζονται σε διάφορα μέρη του πλανήτη μέχρι όλους εκείνους τους ε, ειδικού τεχνολόγους οι οποίοι προστατεύουν τα περίπλοκα δίκτυά μας. Μόλις αυτή την εβδομάδα μπορέσαμε με τον τρόπο αυτό να συλλάβουμε έναν ύποπτο ο οποίος ετοιμαζόταν να φύγει από την χώρα και που είχε κάνει την απόπειρα στο Times Square της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την ικανότητα αυτή. Και γι' αυτό θεωρούμε ότι, θεωρούμε ότι το Terrorist Finance Tracking Program είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει δώσει σημαντική βοήθεια στις προσπάθειες αντιμετώπισης της τρομοκρατίας και από τις δύο πλευρές, από τις δύο του, του Ατλαντικού. Έχει και προβλέψεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Βεβαίω δεν σα μέμφωμαι επειδή αμφισβητείτε ορισμένε πτυχέ του. Το κατανοώ. Μόνο συνεργαζόμενοι θα αντιμετωπίσουμε τι αδυναμίε αυτέ. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα επιτύχουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά εξασφαλίζοντας την προσωπική σφαίρα. Είναι σημαντικό να το πράξουμε αυτό και όσο το δυνατόν συντομότερα. Ως πρώην γερουσιαστή των ΗΠΑ γνωρίζω και πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να καλείται κανεί να κάνει σκληρέ επιλογέ που επιβάλλονται από τι παγκόσμιες προκλήσει προσπαθώντα ταυτόχρονα να τηρήσει τι τοπικέ αξίε. Είμαι βέβαιο ότι όλα αυτά τα περνάτε και εσεί κάθε φορά που κατεβαίνετε υποψήφιοι σε εκλογέ. Όσο περισσότερο έχουμε, περνάμε χρόνο χωρίς συμφωνία για το tracking program που ανέφερα προηγουμένως, τόσο χειρότερα. Ως ηγέτες έχουμε κοινή ευθύνη να πράξουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τα 800 εκατομμύρια ανθρώπων που υπηρετούμε. Έχουμε διαφωνήσει και στο παρελθόν, θα ξαναδιαφωνήσουμε ασφαλώς, αλλά είμαι πεπισμένος επίσης ότι και οι ΗΠΑ και η Ηνωμένη Ευρώπη μπορούν να αντιμετωπίσουν τι προκλήσει του 21ου αιώνα όπω αντιμετώπισαν εκείνε του 20ου αιώνα, εφόσον διαλεγόμαστε ειλικρινώς μεταξύ μας. Κύριε και κύριοι, το θάρρος, μας δίδαξε ο Winston Churchill, είναι αυτό που χρειάζεται για να γύρει κανείς τον άστημά του και να ομιλήσει. Το θάρρος είναι εκείνο που χρειάζεται επίσης για να καθίσει κανείς κάτω και να ακούσει τον άλλο. Βέβαια μέχρι τώρα εγώ μιλώ εδώ. Να είστε βέβαιοι όμως ότι και εγώ και η κυβέρνησή μου και ο πρόεδρός μου έχουμε και πάλι μάθει να ακούμε, να ακούμε τους συμμάχους μας. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Ευρώπη απετέλεσε την πρώτη μου υπερπόντια ε, ε, προορισμό, το πρώτο μου υπερπόντιο προορισμό και του Προέδρου μου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε χρειάζονται την Ευρώπη και με κάθε σεβασμό προς, προς τα πρόσωπά σας θεωρώ ότι και η Ευρώπη χρειάζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα περισσότερο από ποτέ. Θεωρώ λοιπόν την επέτειο τούτης εδώ της εβδομάδος σαν μια καλόδεκτη ευκαιρία για να επανεπιβεβαιώσουμε τα δεσμά των δύο, των δύο λαών μας που έχουμε σφυριλατήσει μέσα από τις φωτιές πολέμων και άλλων ε, ε, δύσκολων περιόδων. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι πρώτα-πρώτα στρέφονται μεν προς τους δε πριν να στραφούν προς οπουδήποτε άλλο για να ζητήσουν την ε, υποστήριξη. Είμαστε, λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι τιμή μας και ε, είμαστε ευγνώμονε που μπορούμε να βαδίσουμε μαζί σας για να αντιμετωπίσουμε τους αγώνες που μας αναμένουν. Ο πρόεδρος Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν υποστηρίζουμε μια ενωμένη, ελεύθερη και ανοιχτή Ευρώπη υποστηρίζουμε αυτά που κάνετε εδώ. Σας ευχόμαστε να σας ευλογεί ο Θεός και να ε, στηρίζει ο Θεός όλες μας τις ε, δυνάμεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Θαυμάσια βάση αποτέλεσε η ομιλία σας για τη μελλοντική συνεργασία, για τις μελλοντικές μας συνομιλίες. Όπως είπατε, να ακούμε ο ένας τον άλλον και να συνεννοούμαστε, να μιλούμε ο ένας τον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τονίσατε αυτό το σημαντικότερο στο οποίο είχαμε καταλήξει και την περασμένη εβδομάδα. Η Ευρώπη χρειάζεται την Αμερική. Να θυμηθούμε τον 20ο αιώνα, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, το σιδηρούν παραπέτασμα. Παραστάτες ε, πολεμούσαμε ένα στο πλευρό του άλλου για να θριαβεύσει η δημοκρατία και η ελευθερία. Και όπως είπατε και εσείς σήμερα χρειάζεται και η Αμερική την Ευρώπη. Ας θυμηθούμε αυτή τη ρίση είναι μια καλή βάση για συνεργασία και εταιρική σχέση. Σας ευχαριστώ και πάλι κύριε Αντιπρόεδρε.